πλαίσια τη νομοθετικής, τακτική νομοθετική διαδικασία, με βάση το άρθρο 78 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου, για πρώτη φορά θα ε, ελέγξουμε το νέο ηλεκτρονικό σύστημα και επίσης θα επικυρώσουμε τη, όλα αυτές τις διαδικασίες με ηλεκτρονική υπογραφή. Διάφορες επιτροπές αποφάσισαν να ξεκινήσουν διαθεσμικές διαπραγματεύσεις